Bien, buenos días. Καλημέρα ξαναλέω ο Πρόεδρος. Είναι 9 ακριβώς. Ε, ε Θα σας πω τα εξή. Έχετε όλη την ηλεκτρονική κάρτα για την ψηφορία, μάλιστα. Και έχετε και τον κατάλογο με την ψηφοφορία, ο καθένας στη δική του, τους συμβασμούς, να μην υπάρχει θέμα πρόβλημα. Έχουμε τα δύο διαδικαστικά για να είναι σαφές ότι ισχύει en el caso de los Όσον αφορά τις καταδιέρεσεις ψηφοφορίας, εάν υπάρχει ισοψηφία, μετράει ότι εγκρίθηκε. Γιατί ο συνήθις κανόν είναι ότι για τις άλλες τροπολογίες, εάν υπάρχει ισοψηφία, ε, θεωρείται ότι απερίφθη. Ενώ για τις συμβαστικές το αντίθετο είναι η διάταξη 209, σύμφωνα σας το λέω, για να είναι σαφές. Κάτι άλλο τώρα. Για τον καφέ. Στις μισή θα έρθει ο καφές. Οπότε ίσως στις μισή με το καφεδάκι ας κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα. Μήπως κάποιος θέλει να βγει για λίγο και να ξαναρθεί μετά από μια μισή ώρα. Επομένως, προχωρούμε. Σπέβδουμε βραδέως, ούτε δεν βιαζόμαστε, αλλά και δεν καθυστερούμε. Ε, γιατί έχουμε αυτό το θέμα τη αλήθεια τη αίθουσα από τη μία μεριά στην άλλη, επομένω με μεγάλη προσοχή α προχωρήσουμε. Για να δούμε τώρα πώ θα προχωρήσουμε, χωρί να υπάρχουν προβλήματα. Και όλοι επομένω α ανοίξουμε τα αυτιά και να δούμε. Α, τι θέλετε, θέλετε κάτι. Έχω ένα συγκεκριμένο θέμα. Ένα διαδικαστικό. Σε σχέση με τρεις τροπολογίες. Να σας τα πω τώρα ή όταν θα έρθει η ώρα στην ψηφοφορία. Yo creo que quizá mejor ahora y así... Καλύτερα τώρα να το πείτε και έτσι να παρακολουθήσουμε όλοι. 4, uh, um, Συμβαστική υπαριθμών 4, 6, και 17. Εδώ έχουμε μια λίστα. Στη λίστα μόνο με του συνδυασμού, αυτά όλα εμφανίζονται ω τροπολογίε. Τροπολογίε όσον αφορά το κείμενο τη Επιτροπή. Βέβαια, σε αυτό αναφέρονται όλε οι τροπολογίε, αλλά σχέση με την τροπολογία υπαριθμών 4, τη συμβαστική αυτή, την 4, την 6 και την 17, ε, το κείμενο αυτής είναι ακριβώς το ίδιο κείμενο, ακριβώς όπως το κείμενο της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να θεωρηθεί η τροπολογία. Πάντως, εγώ αυτό που θα σας πω είναι ότι αυτό μπορεί να θεωρηθεί συμβαστική τροπολογία. Και άρα τα μέλη να μην μπορέσουν να ψηφίσουν τις πραγματικές, αυθεντικές τροπολογίες που εμείς έχουμε κατεβάσει. Ιδίως δε την ε, συμβαστική 17. Και εάν επομένως έχουμε έγκριση της ε, συμβαστικής, τότε η δική μου πρόκειται να καταπέσει. Άρα δεν αποδέχομαι ότι αυτό είναι η ορθή διαδικασία και επομένως θα πρέπει να θεωρηθεί αυτό ως συμβαστική μεταξύ των άλλων συμβαστικών. Αλλά λοιπόν αυτή η εκδοχή δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί η αρχική τροπολογία ως συμβαστική. Και άρα μπορούμε να ψηφίσουμε τις κανονικές τροπολογίες. Λέει ξανά ο εισηγητής. Αυτό ισχύει για το 17, επί της οποίας έχω και εγώ μία. Και θα ήθελα να ψηφίσω επ' αυτής. Δεν είναι πολύ σωστή αυτή η διαδικασία. Εντάξει, να μην δέχεστε τις τροπολογίες του κειμένου της Κομισιόν, αλλά τουλάχιστον να μπορούμε να τις κατεβάσουμε και να περάσουμε από ψηφοφορία ε, ε, ασχέτως και τη απουσία συμβαστικής. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω ότι ισχύει για αυτές τις τρεις περιπτώσεις. Ε, Όντως είναι δύσκολο όταν έχουμε τις συμβαστικές να δούμε τι θα γίνει για να καλύψουμε όλους για τις κανονικές τροπολογίες. Αυτό Κάναμε την τελευταία φορά, προσπάθησα εγώ να το κάνω. Έχουμε το άρθρο 161.3 που λέει εκεί σαφώς ότι ο πρόεδρος μπορεί το βασικό κείμενο να το θέσει πρώτο σε ψηφοφορία ή τις τροπολογίες που πλησιάζουν περισσότερο στο, στην πρώτη στην original εκδοχή και μετά τις άλλες τροπολογίες. Και, και εδώ δεν είναι θέμα προσέγγισης. Ε, είναι ακριβώς ταυτόσιμο. Επομένως έχουμε αυτή την διευκόλυνση από 161.3 και αυτό και το έκανα τότε. Και οπότε στο μέτρο του δυνατού να μπορέσω να προωθήσω όσο γίνεται τους συμβασμούς. Αλλά είναι αδύνατο ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες γιατί πάντοτε υπάρχουν κάποιες τροπολογίες. Οπότε και οι συμβαστικές τροπολογίες δεν καλύπτουν όλες τις αποχρώσεις, όλες τις παραλλαγές. Επομένως με αυτή την ρότα Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις συμβαστικές. Μπορώ να τους ικανοποιήσω όλους, αλλά προσπαθώ να ευνοήσω τις συμβαστικές τροπολογίε. Και τα αυτά τα λέει 161, η διάταξη 161, 3 του κανονού μας. Πρόεδρε, κοιτάξτε, στην τροπολογία 2007, στη σελίδα 127, στο άρθρο 132 ή 32, το απέσυρε. Και εδώ λέει ότι ακόμα είναι προς 120 σελίδα, 127 άρθρο 32 ε, εδώ λέει ότι, ότι, ότι είναι προς ψηφόρια εγώ την έχω αποσύρει είναι η τροπολογία 2007 Σύμφωνα. και αν δούμε πως υπάρξει από αυτού ε, συμβαστική Καντέκ ένα διαδικαστικό θέμα. Μας είπατε πριν ότι στις ψηφοφορίες κατά τμήματα αν υπάρχει ισοψηφία τότε η υπερψήφιση κερδίζει και όχι η καταψήφιση ενώ στην Ολομέλεια γίνεται το αντίθετο. Είστε σίγουροι για αυτό που λέτε. Ναι, ναι, το, το είδαμε, μου το είπαν οι συνεργάτες μας όχι μόνο στην Ολομέλεια, όταν έχουμε καταδιέρεση ψηφοφορία, όταν έχουμε ισοψηφίε στι ε, συμβαστικέ, λέμε ότι εγκρίνεται. Για τι άλλε απορρίπτονται. Αλλά στι καταδιέρεση θεωρούνται εγκεκριμένε. Αυτό μου λένε οι υπάλληλοι, το επιτελείο μα και εγώ του εμπιστεύομαι και το ε, διάβασα και εγώ. Εάν δεν έχουμε κάτι άλλο, επομένω, συνεχίζουμε την ψηφοφορία. Παρακαλώ, προσέξτε όσο μπορείτε περισσότερο και πάμε τώρα στη συμβαστική υπαριθμών 1 αυτή η οποία είναι ε, σπασμένη σε τέσσερα κομμάτια οπότε πάμε στην ε, συμβαστική την πρώτη το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε πέρας Απροβάδο. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτω. Τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Pasamos directamente al compromiso número. Y Και ahora τώρα στην συμβαστική 2. Bueno, yo creo que todos tenemos la misma página. Compromiso número 2. También... Αυτά για το 2. Οπότε τώρα στην και εδώ πέρα έχουμε σε, σε 7 κομμάτια διερημένη. Πρώτο τμήμα, ψηφίζουμε. Τιέρα. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Πέμπτο. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Έκτο. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απροβάδο. Εγκρίνεται. 7, parte 7, comienza. Cierra. Πέρασε. Εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην τροπολογία 655. Σελίδα υπαριθμών 9. 655. βρήκατε, ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα, Envy 21, σελίδα 10. Envy 21. Τι βρήκατε, ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τρία. Και εδώ έχει διαιρεθεί αυτή σε επτά τμήματα. Πρώτη. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρίτο. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Πέμπτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. εγκρίνεται. Έκτο. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Έβδομο. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. NV23. Τι δεν τα 699 στη σελίδα 14. Τη βρήκατε. 699 NV23. Το ίδιο είναι. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτονται. Ή απορρίπτονται και οι δύο. Estamos a la 749. 749, 749 σελίδα 17. 749 του κυρίου Χιούτον ή Χάτον. Ψηφίζουμε. πέρα. Απορρίπτεται. 768. Στην επόμενη σελίδα. 768 Φερέιρα ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται πάμε στην τροπολογία 39 και 783 και NV27 στην ψελίδα 19 ψηφίζουμε πέρας Aprobada. Enmienda 7. 786. Είναι η επόμενη. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 785. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 784. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Aprobada. Enmienda 787. Comienza. Cierra. Πέρασε η επόμενη. Rechazada. Enmienda 788. 788. Πέρασε. Έτσι. Απορρίπτεται. Ρέτζι 38. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Με ισοψηφία. 8-9. 789. Ψηφίζουμε. Τιέρα. Πέρασε. Ρετσαθάδα. Απορρίπτεται. Τα. Comienza. 390 ψηφίζουμε. Πέρας. Aprobada. Envi 28. Comienza. Envi 28. Ψηφίζουμε. Ah, perdón. Está aprobada la 790. Cae 791. Καταπίπτει. Και πάμε στην 791 τέλο 791 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Μισοψηφία. Πάμε τώρα στη συμβαστική αριθμό 4. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στην 800 του κυρίου Σαλαβράκου. Ψηφίζουμε. Δεν λειτουργεί. No, hay dos más del PP. Vamos a seguir como estábamos. Για να, για να δούμε πώς ήταν η κατάσταση. Τι, όχι, όχι, όχι, τίποτα. Άκυρον, άκυρον. Θα το, θα το ξανακάνουμε. Ο, όμως βγήκανε δύο περισσότεροι ψήφοι από το ΕΛΚ και ένας από την ΕΛΔΕ. Για να αρχίσουμε τώρα, ε, ράβε ξύλωνε, καλά, τα πηγαίναμε. Για να δούμε τώρα, δεν δουλεύει το μηχάνημα. Είναι το caso Vamos a repetir la votación. Tranquilidad. Και yo creo que ha Το μηχάνημα φταίει. Πάμε τώρα. Κύριε Ντέβι, κύριε Ντέβι, τι θέλετε, δικαστικό. Ε, ε, το, φωτάκι, ε, όχι, είναι λάθο, φαίνεται. άναψε κατά λάθο φωτάκι. Καλύτερα να με ακούτε, είναι πιο εύκολο αν με ακούτε. Αυτό, αυτό έλεγα κύριε Ντέβης, αλλά δεν με ακούγατε. Έλεγα, φταίει το μηχάνημα και θα το ξανακάνουμε. Οι 800, 800 ψηφίζουμε. No. Όχι, τίποτα. Δεν δουλεύει. No. The machinery doesn't work. No. Yeah, yeah. Yeah, yeah, no, it's, it's, están, están, están funcionando, está la máquina haciéndolo al revés. Yo he puesto negativo, salía positivo. Για να δούμε τι, πώς θα μπορούμε να τη φτιάξουμε, για να προσπαθήσουμε και πάλι. There is a problem with the voting machine. It doesn't accept any. Η μηχανή μου δεν δέχεται τίποτα. Έχω αλλάξει δύο κάρτες και πρέπει να ξαναψηφίσουμε από την αρχή. Δεν το έχω. Δεν το έχω. Το θέμα είναι ότι δεν είναι ότι πετάει την κάρτα, την αποδέχεται, αλλά όταν ψηφίζει το, το αντίστροφο. Το συν το κάνει πλην και αντίστροφος. Το υπέρ κατά και το κατά υπέρ. είναι, είναι, είναι η ώρα, είναι νωρί. Πρωί, πρωί. Τέλος για να ξαναδοκιμάσουμε την 800. No, no, todavía no está puesta. Comienza. Έναρξη ψηφορίας. Ό, τίποτα. No, no funciona. Δεν δουλεύει. Επομένως, τα πράγματα είναι σοβαρά. Bueno, Yo espero que el servicio técnico mira a ver si lo podemos resolver de forma inmediata. no me να δούμε me ames y άμεση no να το λύσουμε. Πάμε καλά. el sistema se ha decantado claramente que no quiere reforma. <laughs> Pero vamos a... Δεν θέλει, δεν θέλει τις αλλαγές το, το μηχανισμό. Δεν του αρέσουν οι αλλαγές, αλλά εμείς θα τις κάνουμε. Bueno, vamos a con humor dentro de todo. Πάνω απ' όλα το χιούμορ. Δεν με νοιάζει εμένα. Αλλά αν ψηφίσουμε μετά σε χειρό, θα γίνουν τα πράγματα πάρα πολύ περίπλοκα. Γιατί έχουμε ψηφοφορίε που ξέρετε που είναι με ισοψηφίες 12, 12 και πέρα και δεν θα μπορούμε να τσεκάρουμε. Θα πρέπει ή να φτιάξουμε το μηχάνημα ή να πάμε αλλού, αλλού που να δουλεύει το μηχάνημα. Δεν γίνεται με τη μέρα της Έχουμε τόσες ψηφοφορίες να ψηφίσουμε και είναι τόσο δύσκολη η ισορροπία. Bueno, si alguien quiere salir, vamos a dar mínimo cinco minutos antes de... Ένα πενταλεπτάκι ε, διάλειμμα και να αρχίσουμε να έρθει ο τεχνικός μου πως το φτιάξει. Break, break. Y espero que sean cinco. Και ελπίζω τα πέντε λεπτά να είναι πέντε λεπτά. Nunca. Ε, El qué, perdón? Vamos a probar a alguien votar lo que sea. Θα δοκιμάσουμε να δούμε αν δουλεύει. Να, να κάνουμε κι εμείς, γιατί κοίταξε είναι αστείο, δεν είναι δύσκολο να κάνουμε αυτά. Από ρελέ. Ε. Van a reiniciar el programa y vamos a ver si hay suerte y... Για να ξεκινήσουμε και πάλι το πρόγραμμα, λέει ο πρόεδρος. Και... Όχι, όχι, όχι, δεν πειράζει. Μην μετά την κουβεντούλα. Δεν θα αρχίσουμε ακόμα την ψηφορία. Για να κάνουμε ακόμα ένα τσεκάρισμα, λέει ο Πρόεδρος. Κάνουμε μόνος ε, μία πλασματική, μία για προπόνηση, μία ψηφοφορία, για δοκιμή. Κάνουμε, τώρα ψηφίζουμε και απαπερίφθη αυτό που σας είπα, αλλά, αλλά δουλεύει. Οπότε συνεχίζουμε αφού ευχαριστήσουμε τους τεχνικούς γιατί τώρα δουλεύει. Και επαναλαμβάνουμε τώρα την 800 τροπολογία, 800 του κυρίου Σαλαβράκου. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 801. Ψηφίζουμε. Α, όχι, όχι. Συγγνώμη, συγγνώμη. Μα, τι, η 890 εγκρίθηκε. Τέλος πάντων. Ένβη 30. Ένβη 30. 30 γιατί είχε, είχε εγκριθεί 790, κατέπεσε 801. Προηγουμένω αυτό είπε ο Πέρασε για την 30. Εγκρίνεται συμβιβαστική 5. Ψηφοφορία. Έναρξη. Όχι, όχι, συμπαθάτε με. Σε δύο τμήματα είναι. Πρώτο τμήμα. 5. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Ένβη 34. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. δεκατρία και 814. Α, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. πάμε στο 811. Η MB31, 811, MB31. 811 και mb 31 Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Είναι ισοψηφία. Τροπολογία 813 και 814. Είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτονται. Συμβαστική 6. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνονται. Τροπολογία 828. Ψηφίζουμε. Πέρας. Ρετσαθάδα. Απορρίπτεται. 42 και μαζί NV36. 42 και MB36. 42 και MB36. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνονται. 8.25. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 8.26. Ψηφίζουμε. Α, όχι. Ε, καταπίπτει αυτή. Η 8.26 καταπίπτει διότι εγκρίθηκε η 7.90. Και πάμε στην 43. 43. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 830 Όστο Οκτώ Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 8.31. Ψηφίζουμε. Πέρασε. 832. τριάντα Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 833. Ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. 8.34. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 8.35. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 8.36. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 8.37. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 44. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 958 και 999 καταπίπτουν διότι εγκρίθηκε 44-838. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Α, όχι. Απορρίπτεται, λέει ο πρόεδρος. 839. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Συμβαστική 7. Ψηφίζουμε. Πέρας. Ε, εγκρίνεται. Και πάμε στην MV38. MV38. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στο 867. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 868 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 871 ψηφίζουμε. Πέρασε. Ε, εγκρίνεται και τώρα πάμε. Χίλια πέντε. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. τριάντα 37. Πέρασε. Απορρίπτεται. 1011 ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. Έμβη 39. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 877. Ψηφίζουμε πέρας. Απορρίπτεται. 878 και 880 που είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνονται. 47. Ψηφίζουμε. Πέρας. εγκρίνεται και πάμε στην 881, 2 και 3 μας. ψηφίζουμε πέρα εγκρίνονται πάμε στην 48 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτωται. 886 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 885 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 884, 7 και έμβη 37 Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στο, στη συμβαστική 9. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. 10 και 11. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνονται. Και πάμε στο 898. Ψηφίζουμε. 898. Φράγα. Στην επόμενη σελίδα. 898. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Το 99. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 993 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 900 και 902 ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 904 και έμβη 42. Ψηφίζουμε πέρας. Απορίτετε. 909 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται 907 ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται 905 ψηφίζουμε πέρας Απορρίπτεται. 906 και 143. 43 Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνονται. 911. 9-11. Ψηφίζουμε. Μισό λεπτό, συγγνώμη. Πάμε στην 908, πατρά. 908 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα την 11. Πέρας. Απορρίπτεται. 9-14. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 9-16. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 9-15. Πέρας. 9, όχι, όχι, λέει πρόεδρος, συγγνώμη, πάμε στο 52. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. MV44. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβαστική 12. <coughs> Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Θα πάμε τώρα στην 13. Ε, Συμβαστική 13. Πέρας. Εγκρίνεται. 14. Πέρασε. Εγκρίνεται. 922, 23 και 24. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 932. και 33. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκλίνεται. Συμβαστική 10 σε τρία τμήματα. Πρώτο. Πέρασε. Εγκλίνεται. Δεύτερο τμήμα. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 945. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 9.46. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται 9.48. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 9.47. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. 9.49. Ψηφίζουν. Πέρασε. Απορρίπτεται. 9.51. Πέρασε. Απορρίπτεται. 9.52, 9.53. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 9.54 και 9.56. Πέρασε. Απορρίπτεται. 9.55 ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. 9.57 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 9.59. Πέρασε. Απορρίπτεται. 9.81. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 9.60 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 9.82. Πέρασε. Απορρίπτεται. Ρέτζι. 42. Πέρασε. 9.90. Με την προφορική που αντικαθιστά το 15 με το νούμερο 12. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε. Έχω αντίρρηση για την προφορική τροπολογία, λέει κυρία Λόβιν. Άρα ψηφίζουμε λόγω της ενστάσεως χωρίς την προφορική. Την ε, ναι, προφορική, ναι. Την 990 χωρίς την προφορική ψηφίζουμε. Πέρας. Γίνεται. 998 ψηφίζουμε. Πέρας. Απολύτωτα. 961. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απολύτωτα. 91. 58, συγγνώμη. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στο 968 πρεσέδο. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 970 ψηφίζουμε. Πέρασε.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 Για να δούμε για την 59, μήπως ε, έχει εγκριθεί κάποια από αυτές από τις οποίες εξαρτάται. No. 59. <clears throat> Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία. 960... Α, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη, γιατί η προηγούμενη εγκρίθηκε. Άρα πάμε στο 971. Ε, ψηφίζουμε, πέρας. Απορρίπτεται. 974. Πέρας. Εγκρίνεται. Και πάμε στο 976. Ψηφίζουμε. Α, όχι, γιατί εγκρίθηκε 974. Α, όχι, λέει ο πρόεδρος. Α, όχι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Πάμε στο 975. Πατράω. 975. Πέρες. Απορρίπτεται. Σε... 276. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 977 και 980. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται και πάμε στο 986 με την 946. 46. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 988. Ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. 985. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 84. Πέρας. Απορρίπτεται. 987 καταπίπτει, γιατί εγκρίθηκε 986 και πάμε στο 1006 ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 2007 ψηφίζουμε. Γίνεται. 994 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 997 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτωτο. Χίλια. Ψηφίζουμε. Απορρίπτωτο. Ενδύ 48. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Χίλια 1003. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 1010 και 49. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 1012 Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνονται. 1013. MV51. 1. Ψηφίζουμε πέρας. Εγκρίνονται. 1014. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτονται. 1015. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 1016. Πέρασε. Απορρίπτεται. Ρέτζε 43 ψηφίζουν. Πέρασε. Απορρίπτεται. 61. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται με ισοψηφία 19. Πέρασε. Για 17. Πέρασε. Απορρίπτεται. 2018. Απορρίπτεται. 52. Πέρας. Απορρίπτεται. 1020. Απορρίπτεται. 53 της ένβη. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 1021. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβαστική 17. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 1030. Φερέιρα. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. MV54. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Τηλεία 29. Εγκρίνεται. 1033. Πέρασε. Απορρίπτεται. 1034. Πέρασε. Απορρίπτεται. 1035. Πέρας. Απόλυτο. 30, 1036. Πέρας. Απόλυτο. 1037. Sí, ¿no? 1037. 1037. ¿Verdad? θάλα. Απορρίπτεται. Και πάμε τώρα στη συμβιβαστική 18. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 19 σε δύο τμήματα. Το πρώτο αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20. σε τέσσερα τμήματα. Πρώτο. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο. Πέρας. Απολύτω. Τέταρτο. Πέρας. Εγκρίνεται πάμε στην συμβιβαστική 21. Στη σελίδα 46. 21. Σε δύο τμήματα. Πρώτο του 21. Πέρασε. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα του 21. Ψηφίζουμε. Πέρας. Α, απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα. Πάμε στη συμβαστική 22. σε δύο τμήματα. Το πρώτο. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Και πάμε στο 23. Σελίδα 50. Σε πέντε τμήματα. Συμβαστική 23. Πρώτο τμήμα του 23. Αρχίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο. Αρχίζει. Ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται τέταρτο. Πέρασε. Εγκρίνεται. Πέμπτο. Πέρασε. Εγκρίνεται. Και τώρα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 Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Περδόν, περδόν. Συγγνώμη, συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Ανοίγει το μικρόφωνο. Πάμε τώρα στην 1227, που είναι προσφύγη. Δεν θα ψηφιζόταν αν είχε απορριφθεί το τμήμα αυτό το δεύτερο του, της συμβαστικής, αλλά εγκρίθηκε και οπότε πάμε τώρα στο 1227. 1227. σελίδα 54. Πρώτα πάμε στο 1227. 1227. Και μετά θα επιστρέψουμε το 24. το 27. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στο 1231. 57 είναι προσθήκη στο 23. 1231-1237. Συμφωνία. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτονται. 24. Τρία τμήματα. Το πρώτο, το 24. Πέρασε. Εγκρίνεται. Δεύτερο. Ούτε το 2 το 3 θα ψηφιστούν. Το τρίτο τμήμα ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε. Cierra. Πέρασε. Απρόβατο. Γίνεται. Πάμε στο 1275 ως προσθήκη. Στο, στη σελίδα 61. 1275. Την έχετε. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβαστική 25. Πέρας. Απορρίπτεται. 25. Και πάμε τώρα στη συμβαστική 26. Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα. Πέρας. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρασε εγκρίνεται. Το τρίτο. Συμβαστική 27. Για να την ψάξουμε. Α, είναι στο 62, σελίδα 62. 27. Και έχει 8 τμήματα. Η 27. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρίτο. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Τέταρτο. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Πέμπτο. Πέρασε. Έκτο. Πέρασε. Απορρίπτεται. Έβδομο. Εγκρίνεται. 8. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 1311 προσθήκη.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 Απορρίφθηκε το 8ο τμήμα. Οπότε τώρα θα ψηφίσουμε 1363 μέχρι 1366 στη σελίδα 70. 1363. Okay. No. Vale. 1360. 1363 ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 64. 1364. Πέρασε. Απορρίπτεται. 1368. Πέρας. Απορρίπτεται. 1367. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 1365 και 66. Πέρας. γίνεται Και πάμε τώρα στο 1311 ως προσθήκη στη συμβαστική 27. 1311. Στη σελίδα 66. Λόβιν, Ρωμέβα και Μπέσε Πέρασε. Απορρίπτωτα. Συμβαστική 28. Σελίδα 71. Συμβαστική 28. Εγκρίνεται. 1387. έως και 91. Πέρασε. Εγκρίνονται. 1386. Απορρίπτεται. 1388. Πέρασε. Απορρίπτεται. Ένδυ 74. Ψηφίζουμε. Πέρασε. απορρίπτεται 1392 και 93 Πέρασε. Εγκρίνεται και πάμε στη συμβαστική 29 και 85 από κοινού. 29 και 85. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνονται. Και πάμε τώρα στη συμβαστική 30. 30. Σε δύο τμήματα. Πρώτο. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Εγκρίνεται. Πάμε στο 1463 ως προσθήκη. 1463, σελίδα 77. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβαστική 31. Συμβαστική 31. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα του 31. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Εγκρίνεται. Συμβαστική 32. Σε πολλά τμήματα. Σε 13 τμήματα. 32. Πρώτο. Πέρας. Ναι, εγκρίνεται. Δεύτερο. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέταρτο. Εγκρίνεται. Πέμπτο. Εγκρίνεται. Έκτο. Απορρίπτωτο. Έβδομο. Έβδομο. Εγκρίνεται. Ναι, ναι. 8. Δεν υπάρχει προφορική τροπολογία. Υπάρχει κάποια αντίρρηση. Ναι. Άρα, αν υπάρχει αντίρρηση, θα ψηφίσουμε την 8η όπως είναι. Το 8ο τμήμα. χωρίς προφορική τροπολογία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Ε, ναι. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. Δέκα. Πέρασε. Έντεκα. Πέρασε. Εγκρίνει. Δώδεκα. Εγκρίνεται. Δεκατρία. ...1562 στη σελίδα 86. Συμβαστική 33. Σελίδα 88. Πέντε τμήματα. Συμβαστική 33 σε πέντε τμήματα. Πρώτο. Ε, εγκρίνεται. Δεύτερο. Πέρασε. Εγκρίνεται. Νομίζω το δεν ψηφίζεται. Πάμε στο 4. Τέταρτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Πέμπτο. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Και πάμε το 1619. 1619. Εγκρίνεται και κατατύπτουν οι επόμενες συμβαστικές και πάμε 1180 στη σελίδα 92 ως προσθήκη στο 33 1180 απορρίπτεται και πάμε στο 34 ψηφίζουμε απορρίπτεται. 35. Ε, Πέρας. Απορρίπτεται. και η 35, άρα θα πρέπει να ψηφίσουμε τις τροπολογίες που περιελάμβανε, που εκάλυπτε η συμβαστική 35. Να τις ψηφίσουμε. MV58 και 1105. Πέρας. Απορρίπτονται.

1269 και 1284. 84 Ψηφίζουμε. ...1666 και NV102. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτονται 1682. 1687. Πέρασε. Απορρίπτεται. 1746. Πέρασε. Απορρίπτεται. 1748 και 105. Ψηφίζουμε. Πέρασε. απορρίπτεται. 1752 ψηφίζουμε. Πέρασε. απορρίπτεται. Και πάμε τώρα στην συμβιβαστική. Στις συμβαστικές μάλλον 36 έως και 45. Από κοινού 36 έως 45. Εγκρίνονται. 39 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα του 39. Το επόμενο του 39. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Δεύτερο τμήμα. Πέρασε. Πάμε τώρα στη συμβιβαστική. 44. Και εδώ είμαστε σε καταδιέρεση, σε τμήματα. Πρώτο. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτω και πάμε. 1781. Σελίδα 106. 1781. Ξεκινάμε. Πέρας. ...1781. Μισό λεφτάκι. Ήρθε ο καφές μεν, αλλά να ψηφίσουμε αυτήν δε. Και μετά διάλειμμα. 1781. Πέρασε. Ρετσαθάδα. 1782. Απορρίπτεται και πάμε στο 1782. Απορρίπτεται. 1783. Απορρίπτεται. Ένβη. 107. Εγκρίνεται. Και 785. Στι 786. Με προφορική τροπολογία, αν δεν υπάρχει ένσταση. Πέρασε. Εγκρίνεται. 788. Εγκρίνεται. Και 787. Απορρίπτωτα. Συμβαστική 46. Πέρασε. Εγκρίνεται. NV108. NV108 πέρασε. Εγκρίνεται. 1793. Ψηφίζουμε. Πέρασε. απορρίπτεται με ισοψηφία 1794 πέρασε εγκρίνεται 1731 απορρίπτεται NV79 Πριν πάμε στο επόμενο κομμάτι της ψηφοφορίας, τι θέλετε κύριε Γκάλαχερ. Θα ήθελα να προσέξετε κάτι. Σε ένα ή δύο τμήματα ψηφίσαμε και αν όχι γιατί. Για ποια μιλάτε. 162. 1602 μάλλον. Την ψηφίσαμε ή όχι. Την ψηφίσαμε. 1602. Σε ποια σελίδα. Δεν την ψηφίσαμε ακόμα γιατί συμπεριλαμβάνεται στο, στη συμβιβαστική 33. Όχι, δεν είναι στη συμβιβαστική. Δεν θα διαβάσω όλο τον κατάλογο εδώ, αλλά έχει τη 1600, 1601, 1602, αλλά όχι τη 1603, η συμβιβαστική 33. ή μάλλον τη 1602. Νόμιζα ότι είναι στο συμβασμό, αλλά βλέπουμε ότι είναι εκεί στο τέλο, στο τέλο, μετά. Οπότε, αν δεν έχετε αντίρρηση, πάμε να ψηφίσουμε την 1602, που ήταν στη σελίδα 90. Λέει ότι περιλαμβάνει στο συμβασμό, αλλά δεν είναι αληθό. Επομένως πάμε να την ψηφίσουμε πέρας. Πέρας. Πέρα. Απορρίπτεται. Mm. Καλώς. Πεντάλεπτο διάλειμμα τώρα. Και μετά θα τον καφέ θα πάμε στο επόμενο τμήμα του ψηφοφορίου.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 Καθίστε παρακαλώ. Ρέγγι 67 Λείπει κανείς. Νομίζω ήρθανε. Η μηχανή δουλεύει, η μηχανή δουλεύει. Λοιπόν, είμαστε όλοι παρόντες. Είμαστε, όχι είμαστε. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε και το δεύτερο μέρος. Λοιπόν. Στο τμήμα 4 υπάρχουν πολλές τροπολογίες. 47, 48, 49, 50, 51, 52 και 93 έχουν καταπέσει. Και γι' αυτό θα ψηφίσουμε τώρα την περίφ 67. Περίφ 67 αρχίζει. 108 Είπα ότι οι συμβιβαστικές 47 με 53 έχουν γίνει ή καταπέσει. Λοιπόν, είναι μετά από αυτές. Λοιπόν, Ρέγγι 67 ψηφίζουμε. Έληξε. Εγκρίνεται. Τώρα Η συμβιβαστική 54. Στη σελίδα 128. Μην εξάπτεστε, λοιπόν. Υπάρχει συμβιβαστική 54 σε τέσσερα τμήματα. Τέσσερα. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Έλξε. Έληξε, είπα. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Α. Α ναι. Όχι, όχι. Έχει καταπέσει, έχει καταπέσει. Συμβιβαστική 55 τώρα, τα άλλα τμήματα έχουν καταπέσει λέει. ...1797. 1797 ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. Καθώς και οι 2000, τώρα οι 2020. Η τελευταία από αυτό το τμήμα εδώ. Ψηφίζουμε 2020. Έλξε. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 55 σε 5 τμήματα. 55 σε 5 τμήματα. Πρώτο τμήμα. Έλεξε. 55 Δεύτερο τμήμα. εγκρίνεται τρίτο τμήμα ισοψηφία απορρίπτεται α όχι είπαμε ότι ε, αυτή την περίπτωση εγκρίνεται στις κατατμήματα τέταρτο τμήμα εγκρίνεται πέμπτο τμήμα ισοψηφία εγκρίνεται δύο χιλιάδες πενήντα στη σελίδα 133. 133 2059 που προστίθεται στη συμβιβαστική 55 λοιπόν αρχίζει η ψηφοφορία ξε Πορύπτεται. συμβιβαστική 56 εγκρίνεται. Συμβιβαστική 57. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 58 στη σελίδα 136. Συμβιβαστική 58 αρχίζει η ψηφοφορία. Okay. εγκρίνεται. Τώρα η συμβιβαστική 59. εγκρίνεται. 2098 προστίθεται στην 59. εγκρίνεται. Τώρα η 2106. Α, όχι, καταπίπτει, καταπίπτει. NV 132. NV 132. Εγκρίνεται.

Απορρίπτεται 208. Απορρίπτεται 209. Απορρίπτεται 210. Απορρίπτεται 211. απορρίπτεται 212 ε, αρχίζει απορρίπτεται NV 134 εγκρίνεται 213 Απορρίπτεται. 214. Απορρίπτεται. 215. Εκεί. ερμά Απορρίπτεται. 216.

εγκρίνεται. NV 135 εγκρίνεται NV 136 εγκρίνεται NV 137

Συγκρινέται 224 224 απορρίπτεται 222 απορρίπτεται

εγκρίνεται. 227. Απορρίπτεται. 228. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 60.

του κυρίου Αρσένη. Απορρίπτεται. NV 140. Απορρίπτεται. 240. απορρίπτεται 242 απορρίπτεται 243 απορρίπτεται NV εγκρίνεται 2.146. Πορύπτεται 2.145. εγκρίνεται συμβιβαστική 62 εγκρίνεται συμβιβαστική 63 εγκρίνεται συμβιβαστική 64 εγκρίνεται Δύο 2.161 εγκρίνεται 2.162 εγκρίνεται επόμενη ομάδα Συμβιβαστική 65. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 66. 6. Εγκρίνεται. 2.191 2.191 εντάξει ως προσθήκη στη συμβιβαστική 65 εγκρίνεται συμβιβαστική 67 Υπάρχει και μια προφορική τροποποίηση εδώ. Είναι κανείς ακατά, Όχι. Μαζί με την προφορική λοιπόν. Μαζί με την προφορική. Το αρχικό κείμενο πρώτα, ε, το αρχικό κείμενο, συγγνώμη. Το αρχικό κείμενο ψηφίζουμε. να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Το αρχικό κείμενο της συμβιβαστικής τροπολογίας 67. εγκρίνεται. Και τώρα η προφορική τροποποίηση στον στη συμβιβαστική 67 είναι κανείς κατά, όχι,

Κλείνει, απορρίπτεται. 2.201. Ανοίγει η ψηφοφορία. Κλείνει. Εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στο 196. Εκατόν ενενήντα έξι. Αρχίζει η ψηφοφορία, κλείνει. Απορρίπτεται. 2202, 2202. Κλείνει. Απορρίπτεται. 2203. Αρχίζει. Κλείνει. Εγκρίνεται. 2204. Αρχίζει. Κλείνει. εγκρίνεται. Ενδύει 148. Ανοίγει, κλείνει. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 68. 68 σε δύο σκέλη. Πρώτο σκέλος, αρχίζει η ψηφοφορία. Κλείνει. Εγκρίνεται. Και το δεύτερο σκέλος, αρχίζει η ψηφοφορία. Κλείνει. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 69 που αποτελείται από τέσσερα μέρη το πρώτο μέρος. Αρχίζει η ψηφοφορία για το πρώτο μέρος. Κλείνει. Συμβασμό 69, πρώτο μέρος. μέρο. 148 150 όλα. Συμβασμό 69, πρώτο μέρος, αρχίζει η ψηφοφορία, κλείνει. ψηφίζουμε τώρα για το πρώτο μέρος του Συμβασμού 69. Εντάξει. Αρχίζει η ψηφοφορία. Είστε έτοιμοι. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Αρχίζει η ψηφοφορία. Με συγχωρείτε, υπάρχει μία προφορική τροπολογία αν δεν έχετε αντίρρηση. Εδώ πέρα αρχίζει η ψηφοφορία, κλείνει, εγκρίνεται. Τρίτο μέρος. Tierra. Aprobada. Cuarta parte, también con una enmienda λοιπόν. oral. Si nadie se... Λοιπόν, έχουμε και την... Ε, συμπεριλαμβάνεται και η προφορική τροπολογία. Υπάρχουν ε, ε, αντιρρήσεις, αλλά όχι προφορική τροπολογία, από ό,τι βλέπω. Το τέταρτο μέρος ήταν η προφορική τροπολογία. Εφόσον όμως δεν υπάρχει προφορική τροπολογία, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. No se vota. Eh, pasamos al compromiso 70. Compromiso 70. Comienza. 70. Ερχόμαστε στο COMP 70, συμβιβασμό 70. Αρχι, αρχίζει, κλείνει, εγκρίνεται. Το 71 αρχίζει η ψηφοφορία κλείνει. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22-21 αρχίζει. 2221. 22-21. Αρχίζει η ψηφοφορία, κλείνει. Εγκρίνεται. 22-19 αρχίζει, κλείνει. Απορρίπτεται. 22-22. Αρχίζει, κλείνει. Εγκρίνεται. 22-20. Αρχίζει. Κλείνει. Απορρίπτεται. 22-25. Κλείνει. Απορρίπτεται. Ερχόμαστε τώρα στην τροπολογία NV149. Ανοίγει κλείνει. Εγκρίνεται. Δεύε 12 αρχή ψηφοφορία. Το ΔΕΒΕ 12. Εντάξει, αρχίζει η ψηφοφορία, κλείνει. Εγκρίνεται. Ερχόμαστε στην τροπολογία 2231. Κλείνει. Εγκρίνεται. 201. 201. Αρχίζει. Κλείνει. Απορρίπτεται. 2232. Όχι, με συγχωρείτε. Όχι. Το DEV 12 εγκρίθηκε. Με συγχωρείτε. Ερχόμαστε στο 22.35. Αρχίζει. Κλείνει. Απορρίπτεται. 22.38. Όχι, με συγχωρείτε. Θα γυρίσω πίσω, διότι, διότι ξέχασα την τροπολογία NV150 πιο ψηλά. Αρχίζει. Ψηφοφορία, κλείνει. Απορρίπτεται. Το 2236. ΔΕΒΕ 15. Απορρίπτεται. 22.37. Αρχίζει, κλείνει, Ψηφορία. Απορρίπτεται. Τώρα είμαστε στο 22.38. Αρχίζει, κλείνει. Απορρίπτεται. 22.39. κλείνει, εγκρίνεται. 22.40 κλείνει, απορρίπτεται. 22.41 κλείνει, εγκρίνεται. 22.42 ανοίγει, κλείνει. Απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 16. Κλείνει. Εγκρίνεται. 22.43. Αρχίζει η ψηφοφορία. Κλείνει. Απορρίπτεται. 22.45. Αρχίζει. Κλείνει. Απορρίπτεται. Δεύε 17. Αρχίζει. Κλείνει. Απορρίπτεται. 22.47. Αρχίζει. Κλείνει. Γυ, γυρνάμε πίσω. Το DEV 17 εγκρίθηκε. Το Ένβι 151. Αρχίζει η ψηφοφορία εδώ. Για το Ένβι 151. Κλείνει. Απορρίπτεται. 22.47. Αρχίζει. Κλείνει. Απορρίπτεται. 22.48. Αρχίζει. Κλείνει. Απορρίπτεται. Ερχόμαστε τώρα στο συμβιβασμό 72, κομπ 72. Αρχίζει ψηφοφορία. Κλείνει. Εγκρίνεται. Συμβασμός 73, κομπ 73. Αρχίζει η ψηφοφορία. Κλείνει. Εγκρίνεται. συμβιβασμό 74, κόμπε 74. Αρχίζει. Στην ίδια σελίδα, 154 πάντοτε. Το κόμπε 74 αρχίζει η ψηφοφορία, κλείνει. Εγκρίνεται. 2260. Αρχίζει η πληροφορία. Κλείνει. Απορρίπτεται. 2.310. το 2310 σελίδα 159 προς τα κάτω με παχιά γράμματα 2310 σελίδα 159 αρχίζει η ψηφοφορία κλείνει απορρίπτεται 2311 αρχίζει κλείνει εγκρίνεται. 23.12 αρχίζει. Κλείνει. Απορρίπτεται. Ένβη 155 αρχίζει. φορια Κλείνει. Εγκρίνεται. 23-13 και 23-14. Αρχίζει η ψηφοφορία. Κλείνει. Απορρίπτεται. 23-16 αρχίζει. Κλείνει. Απορρίπτεται. 208 αρχίζει. Κλείνει. εγκρίνεται. 23.15 αρχίζει, κλείνει, απορρίπτεται. 23.18 αρχίζει, κλείνει. Απορρίπτεται. 23.19 Αρχίζει, κλείνει. Απορρίπτεται. 23, 20, 21 και 22. Κλείνει. Απορρίπτεται. 23, 23 και 23-42 αρχίζει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 23-24 αρχίζει. Κλείνει. Εγκρίνεται. 23-25 αρχίζει. Κλείνει. Απορρίπτεται. 23-26 αρχίζει, κλείνει. Απορρίπτεται. 23-27 αρχίζει, κλείνει. Απορρίπτεται. 23-28 αρχίζει, κλείνει. Απορρίπτεται. Envy 155. Αρχίζει. Εγκρίνεται. 23-29. Αρχίζει. Κλείνει. Εγκρίνεται. 23-30. Κλείνει. Απορρίπτεται. Ένβη 155. Αρχίζει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 2331. Απορρίπτεται λέει ο πρόεδρος. 2.732. Απορρίπτεται. Με ισοψηφία. 2734, Πέρας. Απορρίπτεται. 2.338. Πέρασε. Εγκρίνεται. 2.337. Δίκαια στο 39. Απορρίπτεται. 2.340. Απορρίπτεται. 1.435. Απορρίπτεται. NV 155. Απορρίπτεται. 2000. 341. Ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. 2343. Απορρίπτεται. 1744. απορρίπτονται. 2.000... Ε, συγγνώμη, 210. Απορρίπτονται... Πύλες 352 και 53. Απορρίπτονται. Και πάμε τώρα το 1754. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 1359. Ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. 1760. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.356 απορρίπτεται

εγκρίνεται 2363 2.764, 2.763 εγκρίθηκε, 2.764, αχ, συγγνώμη, συγγνώμη, 2.370 Πέρας. Α, απορρίπτεται. 2369. Απορρίπτεται. 2365. Απορρίπτεται. 2368.

καταπίπτει 2773 απορρίπτωτο NV 156 πέρας εγκρίνεται 2374

Πέρασε. Απορρίπτεται. 2.400. Το οκτώ. πέρασε. Εγκρίνεται. Και πάμε στο 2799. εγκρίνεται. 2401. Βιβλία 402. Εγκρίθηκε η 401. Βιβλία 403. Απορρίπτεται. 213. Πέρασε. Εγκρίνεται. 2404. Δύο 1406 Εγκρίνεται. Συμβαστική 76. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2414. 313. Πέρασε. Απορρίπτεται. 2315. Πέρασε. Απορρίπτεται. 2316. Πέρασε. απορρίπτεται 1418. απορρίπτεται 1417 πέρασε απορρίπτεται συμβαστική 77 σε δύο τμήματα το πρώτο Πέρασε. Εγκρίνεται. Δεύτερο. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 78. Πέρασε. Εγκρίνεται. 79. Πρώτο τμήμα του 79. Δεύτερο. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Απορρίπτεται. Και πάμε... Εσύ όχι. Πρέπει να πάμε στην 2439. Ε, γιατί στο τρίτο τμήμα είχαμε απόρριψη. 2.439 τώρα. Συμφωνεί. Ψηφίζουμε. Πέρας, απορρίπτεται. Έμβη. 159. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 214. Εγκρίνεται. 2.440. Απορρίπτεται. Και 2.441 ψηφίζουν. Πέρασε. Απορρίπτεται. Πάμε τώρα στη συμβαστική 80. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 81. Οδόντα εγκρίνεται. 83. Σε δύο τμήματα. Το πρώτο. Πέρασε, εγκρίνεται. Το δεύτερο. Εγκρίνεται. τέσσερα. 84 que también está dividido Σε έξι τμήματα. Συμβαστική 84. Πρώτο τμήμα. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Είναι προφορική τροπολογία, αλλά δεν είναι αποδεκτή. Άρα δεν θα ψηφιστεί. Και πάμε στο τρίτο τμήμα. Ψηφίζουμε το τρίτο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα. Με προφορική τροπολογία. Όχι. Δεν τη θέλετε και άρα δεν θα γίνει ψηφορία για το τέταρτο τμήμα. Πέμπτο. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε, πέρας. Εγκρίνεται. Έκτο. Ψηφίζουμε. Se cierra. Aprobada también. Εγκρίνεται και αυτή. Και πάμε εγώ τώρα. Πού, πω 82. Μία δέσμη συμβαστικών διατάξεων 82 με την 87 και την 75. Οπότε ε, και εδώ έχουμε ει τμήματα. Τέσσερα. Πρώτο. Εγκρίνεται. Δεύτερο. Εγκρίνεται το δεύτερο, πάμε στο τρίτο. Ψηφίζουμε, πέρας. Εγκρίνεται. Τέταρτο. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. Πάμε στο τροπολογία 2534. Δύο, πέντε, τρία, τέσσερα. Το βρήκατε. Στο 2534 είμαστε. Ναι, το βρήκατε. Απορρίπτω. Συμβαστική 86. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 2... 224. Ναι. 2, 2, 4. Αλλά μαζί δείχνετε 67, 38 και 39. Ψηφίζουμε. Πάμε σε προφορική τροπολογία που έρχεται από τους σοσιαλιστάς. Αφού δεν αποδεικτεί δεν θα την ψηφίσουμε και πάμε στο 2545. 2545. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 2540. Όχι, 2535 διορθώνει. 2535. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 2.542 και 226. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. 228. Ya está. Pasamos a los, al 228, el último bloque. Venga. 228. <clears throat> Hay una enmienda oral también del señor Cadet. ¿Alguien se opone? Υπάρχει προφορική τροπολογία του ΚΑΝΤΕ και έχετε ένσταση. Όχι, αλλά πάμε στο 228 που είναι προφορική. Πέρας. Απροβάδα. Πασάμος a los recitals. Eh, 231. Comienza. Cierra. Πέρας. Rechazado. Enmienda 1. Comienza. Η 1, υπαριθμόν 1, ναι, πέρας. Εγκρίνεται. 200, πόσο, πόσο, πόσο, 2.34, μαζί με την ένβη 3. Ε, ψηφίζουμε, πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 88. Ψηφίζουμε. Γίνεται. 239. Προσθήκη στο 88. 239. Κύριε Χάντον. 239. Απορρίπτωτο. Ρέχει, ρέτζι, τρία. απορρίπτεται. 243. Απορρίπτεται. 244. Απορρίπτεται.

απορρίπτωτο. Ρέτζε τέσσερα. ψηφίζουμε. Οδόντα εννέα. ¿eh? Eh, όχι, δεν έχουμε εδώ κατά τμήματα. Όλοι μαζί οι 89. Εγκρίνεται. Πάμε στο 90. Και εδώ το ίδιο, στο σύνολό της. Comienza. Ψηφίζουμε το 90. Πέρασε. καταπίπτει γιατί δεν εγκρίθηκε 25 ή 34. Καταπίπτει το 91 και πάμε στο 92. 92. σε δύο τμήματα. Το πρώτο. δεύτερο. Εγκρίθηκε το πρώτο, εγκρίθηκε το δεύτερο και πάμε στο Ρέτζι 5. Απορρίπτεται. Τέσσερα. Πέρασε. Εγκρίνεται 266. Πέρασε. Εγκρίνεται 267. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Ε, συμβιβαστική 94. Πέρας. Εγκρίνεται. 270. Απορρίπτεται. 95. εγκρίνεται 275 πέρασε απορρίπτεται 276 πέρασε Ένβη. 6. Ψηφίζουμε ε, πέρας, εγκρίνεται. 277. Πέρας. Απορρίπτεται. 278. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 96. Πρώτο τμήμα. Εγκρίνεται. Αν μπορείτε το δεύτερο τμήμα. Α, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Έχει κάνει λάθο ο πρόεδρο, διορθώνει. Και πάμε στο 294. 2-9-4. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 297. Πέρασε. Εγκρίνεται. 287 εγκρίνεται και πάμε στο 2. Όχι, όχι. Λέω πρόεδρος. Πάμε στο 292. 292 ψηφίζουμε. Απορρίπτεται. 686. Δύσκολα. Απορρίπτεται. 288. Απορρίπτεται. 290. Εγκρίνεται. 289. Απορρίπτεται. 293.

απορρίπτεται 301 πέρας απορρίπτεται 300 πέρας εγκρίνεται 5 mm. 299 ως προσθήκη. Πέρας. Απορρίπτεται. 298. Πέρας. Απορρίπτεται. 5. Πέρας. απορριπτεται πρωτα πρώτα θα ψηφίσουμε την 302 πριν την 303. Απορρίπτεται.

Απορρίπτεται. 307. Απορρίπτεται. 6 με την 305. Εγκρίνεται 308. Όχι, πάμε στο 309. Απορρίπτεται, 306. Απορρίπτεται, 311. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. 312. Πέρασε. Απορρίπτεται. Ρέτζε. 10. Απορρίπτεται. 313. Πέρας. Απορρίπτωται. Καταπίπτει. Τα 316. 310. Πάμε στο 316. Απορρίπτεται. 218. Rechazada. 300 φως, 317 φως, 320. 320 και 21. Τέλος. Απορρίπτονται. Ρέτζι 12 απορρίπτεται 324 πέρας Γίνεται Ρέτζι 13. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 327. Απορρίπτεται. NV8. Απορρίπτεται. 326 και 329. Κρίνονται. 328. Συμβαστική 97.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 Τροπολογία 359. Πέρασε. Απορρίπτεται. 362. Δύσκολα. Απορρίπτεται 364.

Ορίπτεται. 363. Γκρίνεται. Περίφ 9. Περίφ 9. Όχι. Α. Ε, ε, 11. Απολογία 11. Η ισοψηφία εγκρίνεται. Απορρίπτεται λέει ο πρόεδρος. 12. Απορρίπτεται. 12. 12. Εγκρίνεται. 367. Απορρίπτεται. 368. Εγκρίνεται. 371. Απορρίπτεται. 372. Απορρίπτεται η ισοψηφία. 373. Απορρίπτεται. 369. που ορίπτεται. 370 ως προσθήκη. Γίνεται 10 Τρία, εφτά, τέσσερα. Απορρίπτεται. 375. Απορρίπτεται. NV11.

απορρίπτεται. 387 εγκρίνεται 382 εγκρίνεται 384 που ορίπτεται. Τριακόσια ογδόντα εννέα. Εγκρίνεται. Τριακόσια ενενήντα. απορρίπτεται 391 απορρίπτεται 392 απορρίπτεται

395, 96, 97, 98, 99, 400 και 401. εγκρίνονται συμβιβαστική 101 101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

445. Απορρίπτεται. Ρέγγι 20. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 102. Εγκρίνεται. 17. Απορρίπτεται.

απορρίπτεται 462 και 469 εγκρίνονται 465 εγκρίνεται 468

απορρίπτεται 476 εγκρίνεται 479 εγκρίνεται 472 απορρίπτεται 474 εγκρίνεται 478. όχι ε, δεν αγορά ε. όχι 482 ε, μήπως

Κλείνει. Απορρίπτεται. 483. Ανοίγει, κλείνει. Εγκρίνεται. 484 αρχίζει, κλείνει. Απορρίπτεται. 485 Αρχίζει, κλείνει. Απορρίπτεται. ένδυ 16 αρχίζει. Κλείνει. Εγκρίνεται. ΡΕΓΚΙ 23 αρχίζει. Κλείνει. Εγκρίνεται. Δεύε 1. Αρχίζει. Κλείνει. Απορρίπτεται. 487 αρχίζει, κλείνει. Απορρίπτεται. 488 αρχίζει, κλείνει. Εγκρίνεται. 489. Αρχίζει. Κλείνει. Απορρίπτεται. 490. Αρχίζει η φοβολία, Κλείνει. Εγκρίνεται. 491. Αρχίζει. Κλείνει. Απορρίπτεται. n 17. Καταπίπτει. Ρέγγι 24. Αρχίζει η ψηφοφορία. Κλείνει. Απορρίπτεται. Ρέγγι 25. Αρχίζει. Κλείνει. Απορρίπτεται. 4-9-2 αρχίζει. Κλείνει. Απορρίπτεται. 4-9-3-4-9-4 αρχίζει. Κλείνει. Απορρίπτεται. 4-9-5 ανοίγει. Αρχίζει. Κλείνει. Απορρίπτεται. 4-9-6. 498. Αρχίζει, κλείνει. Απορρίπτεται. 499. Αρχίζει, κλείνει. Απορρίπτεται. 496. Αρχίζει η ψηφοφορία, κλείνει. Απορρίπτεται. 4-9-7 αρχίζει αρχίζει, κλείνει. Απορρίπτεται. Το 19. Αρχίζει η ψηφοφορία, κλείνει. Απορρίπτεται. 501 αρχίζει, κλείνει, απορρίπτεται. 500 αρχίζει, κλείνει, απορρίπτεται. Ρέγγι 26 αρχίζει, κλείνει, απορρίπτεται. 502 αρχίζει, Κλείνει. Απορρίπτεται. 503. Αρχίζει. Κλείνει. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 103. Κομπ 103. Αρχίζει. Κλείνει. εγκρίνεται. Ερχόμαστε στο 509. 509 αρχίζει, κλείνει. Απορρίπτεται. 511 αρχίζει, κλείνει. Απορρίπτεται. 512 αρχίζει, κλείνει. απορρίπτεται. 514 αρχίζει, κλείνει. Απορρίπτεται. 513 αρχίζει, κλείνει. Απορρίπτεται. 515 αρχίζει, κλείνει. απορρίπτεται. 5.17 αρχίζει, κλείνει. Απορρίπτεται. 5.16 αρχίζει, κλείνει. Απορρίπτεται. 5.18 αρχίζει, κλείνει. Εγκρίνεται. 5.19 αρχίζει, κλείνει. Απορρίπτεται. Ρέγγι 27 αρχίζει. Κλείνει. Απορρίπτεται. 524 αρχίζει. Κλείνει. Απορρίπτεται. Ισοψηφία. 522 αρχίζει. Κλείνει. απορριπτεται 5.20. αρχίζει. Κλείνει. 5.25. Αρχίζει. Κλείνει. 5.25. Εγκρίνεται. Ωραία. 5.23. Αρχίζει. Κλείνει. Εγκρίνεται. 5.21. Αρχίζει. Κλείνει. Απορρίπτεται. 5.26. Αρχίζει. Κλείνει. Απορρίπτεται. Ρέγγι 28 αρχίζει. Κλείνει. Απορρίπτεται. 527 αρχίζει. Κλείνει. Εγκρίνεται. 528 αρχίζει. Κλείνει. εγκρίνεται. 529, 530 και 531, τα τρία μαζί. Αρχίζει η ψηφοφορία. Κλείνει. Απορρίπτεται. 533. Αρχίζει, κλείνει. Απορρίπτεται. 537. 537. Αρχίζει, κλείνει. Απορρίπτεται. 538 αρχίζει. Κλείνει. Απορρίπτεται. 539 αρχίζει. Κλείνει. εγκρίνεται. 5.40. 5.40. Αρχίζει, κλείνει. Απορρίπτεται. 5.41. Αρχίζει. Απορρίπτεται. 21. Αρχίζει, κλείνει. εγκρίνεται. 5.42 αρχίζει, κλείνει. Απορρίπτεται. 543 αρχίζει, κλείνει. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22 αρχίζει, κλείνει. Απορρίπτεται. 5.45 αρχίζει, κλείνει. Απορρίπτεται. 5.46 αρχίζει, κλείνει. Εγκρίνεται. 5.47 αρχίζει, κλείνει. Απορρίπτεται. 5.49. 5.49 αρχίζει. Κλείνει. Απορρίπτεται και πάμε στο 150. Απορρίπτεται. Και πάμε στην συμβαστική 104 εις δύο τμήματα. Το πρώτο εγκρίνεται. Δεύτερο πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε στην 24.

απορρίπτεται 567 απορρίπτεται 568 569

Ωραία και τώρα. Τελειώσαμε. Αλλά απομένει να ψηφίσουμε την νομοθετική πρόταση όπως τροποποιήθηκε. Επίσης, είπαμε να υπάρξει κάποιο χρονικό περιθώριο, αλλά τώρα όμως δεν το έχουμε γιατί είμαστε 12.30. Ε, πάντως συγχαρητήρια σε όλους. Ήταν ε, πάρα πολύ άρτια η διαδικασία, δείξαμε ευελιξία κλπ. Οπότε Πάμε στις 3 τώρα. Στις 3 θα ξανάρθουμε. Βέβαια στις 4 θα συνεχίσει η Επιτροπή επομένως. Θα πρέπει να είμαστε εδώ όλοι στις 3 και να μην αργήσουμε για να κάνουμε απλώς την ψηφοφορία της, ε, την υπόλοιπη ό,τι μένει, δηλαδή το σύνολο του, του νομοθετικού κειμένου. Κάποιοι ζητήσει το λόγο, αλλά τέλος πάντων... Α, ο κύριος Ντέιβις. Ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για όλη τη δουλειά της στην κατάρτιση αυτού του πολύπλοκου καταλόγου ψηφοφορίας και για τον τρόπο με τον οποίο διευθύνεται την συνεδρίαση. Αλλά γιατί να μην ψηφίσουμε τώρα και να περιμένουμε το απόγευμα. Bien. Eh, hay dos, Sí, Antinoro. Scusi eh, Πρόεδρε, αν χρειαστεί μισή ώρα για να είναι όλα εντάξει, τότε εντάξει, καταλαβαίνω, αλλά να ψηφίσουμε στις τρεις γιατί, για ποιο λόγο, γιατί μεταθέτουμε την ψηφοφορία. Να σας απαντήσω μεταξύ άλλων. Γιατί και από τις 3 προβλεπόταν ψηφοφορία, όμως στα τελειώσαμε στις 12.30. Για ρίξτε μια μετιά στην ημέρα σε διάταξη. Μην μου λέτε όχι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Και μετά θα τα βρούμε. Να κάνουμε ό,τι θέλετε, αλλά μην μου λέτε όχι, γιατί στη μερισσία διάταξη λέει ότι από τις 9 μέχρι τις 12.30 ψηφοφορία αλλά και από τις 3 από τις 3 και μετά Μη μου λέτε όχι πέστε μου έκανα λάθος ή δεν το βλέπω Μη μου λέτε όχι τέλος πάντων αυτή είναι η πρόταση να συνεχίσουμε την ψηφορία και επίσης υπάρχει κάποια ομάδα η οποία είχε ζητήσει να γίνει ένα διάλειμμα 15 ως 20 λεπτών μέχρι την τελική ψηφοφορία. Όμω τώρα έχουμε ξεπεράσει το όριο τη πρωινή συνεδρίαση. Και το φυσιολογικό είναι να γίνει αυτό που σα είπα. Τώρα, εάν όλοι μαζί, ομοφόνο, θέλετε τώρα να ψηφίσουμε, να ψηφίσουμε. Μόνο αν υπάρχει ε, ομοφωνία. Αλλιώ θα κάνετε αυτό που λέει ο πρόεδρο, ο οποίο διευθύνει τη διαδικασία. Θέλουν όλοι τώρα να γίνει ψηφοφορία. Όχι. Άρα θα συνεχίσουμε την ψηφοφορία στι 3. 3. Και μετά θα συνεχιστεί η συνεδρίαση της ε, Επιτροπής. Sí, señora Rodus. Señora Rodus tiene γνωρίζετε, παρακολούθησα πολύ προσεκτικά αυτή τη ψηφοφορία και έχω την εντύπωση ότι υπάρχει σχεδόν ομοφωνία θα έλεγα. Λοιπόν δεν πρέπει να υπάρξει μια παύση τώρα. Δεν ξέρω τι πιστεύετε. Νομίζω δεν χρειάζεται να, να γίνει διακοπή. Θα μπορούσαμε να κάνουμε τώρα την οριστική ψηφοφορία. Εάν κάποιο θέλει διακοπή, τότε τα πράγματα είναι πλέον καθαρά. Θα διακόψουμε. Αν όμω όλοι οι παρόντε και οι παρούσε ε, συμφωνούν, μπορούμε να κάνουμε τώρα την τελική ψηφοφορία. Señora Patrao. Eh, nós tínhamos anteriormente pensado em ε, είχαμε σκεφτεί το εξή ε, Να υπάρξει μια διακοπή προκειμένου να αξιολογήσουμε τα πράγματα. Έχουμε εδώ ε, μπροστά μας 211 σελίδες δεν ξέρω αν όλοι ε, ε, έχουν καθαρό μυαλό ακριβώς. Και δεν καταλαβαίνω γιατί ένα τόσο σημαντικό έγγραφο, το οποίο σε μεγάλο βαθμό θα καθορίσει την κοινή αλληλευτική πολιτική μέχρι το 2020, ε, δεν αξίζει να έχει λίγο χρόνο, να το σκεφτούμε δηλαδή ώστε να μπορούμε να ψηφίσουμε ήρεμα και κατά συνείδηση. Διότι αν λέει η Μεσαία Διάταξη ότι μπορούμε θα ψηφίσουμε στις 3, τότε